dear colleagues, uh, three past nine, let's start. Συνάδελφοι, είναι 9 και 3, οπότε ας ξεκινήσουμε. Καλημέρα σε όλους. Νομίζω πως έχετε όλοι λάβει την ημερήσια διάταξη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο αίτημα για τροποποίησή της. Εάν όχι, θεωρούμε πως εγκρίνεται. Περνάμε στο σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων και συγκεκριμένα των πρακτικών της συνεδρίασης Τη Δευτέρα και 3 Σεπτεμβρίου. Έχετε λάβει το σχετικό έγγραφο των πρακτικών. Εάν λοιπόν δεν υπάρχουν αντιρρήσει ε, που θα πρέπει να εκφραστούν έως τα τέλη της σημερινής ε, συνεδρίασης, ε, θα θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί. Μετά, επόμενο σημείο είναι οι ανακοινώσεις μου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές. Και εδώ πάλι έχετε λάβει το σχετικό έγγραφο όπω εκείνο των πρακτικών της προηγούμενη συνεδρίασης, οπότε αν δεν υπάρξουν και πάλι αντιρρήσει σε σχέση με τα λόγω έγγραφα και τα πρακτικά της συνεδρίασης των συντονιστών θεωρούνται ως εγκεκριμένα. Περνάμε στο σημείο 5, ανακοινώσει του Προέδρου. Ως συνήθως έχουμε web streaming και σήμερα τη σημερινή συνεδρίαση, οπότε σίγουρα έχουμε πολλούς τηλεθεατέ από το Λουξεμβουργό ως το Λούνεμπουργκ και από το Ταλίν έως τη Θεσσαλονίκη που μας παρακολουθούν, οπότε τους καλωσορίζω όλους. Και έχουμε πέραν του web streaming και διερμηνία, οπότε για να σας προλαβαίνουν οι διερμηνείς να μιλάτε αργά, να μιλάτε καθαρά και φροντίστε να εμφανίζεστε στην οθόνη και να μιλάτε με καθαρή φωνή έτσι ώστε να μπορούν οι διερμηνείς να σας μεταφράζουν. Αυτά λοιπόν ως προς τις ε, ανακοινώσεις από την δική μου πλευρά και από εκεί και μετά μια πιο ασυνήθιστη ανακοίνωση είναι η ακρόαση που θα λάβει η χώρα σε ό,τι αφορά ε, τον επίτροπο που έχει επιλεγεί, τον Φιλ Χόγκαν δηλαδή, για τα ζητήματα εμπορίου. Την Δευτέρα λοιπόν, 30 Σεπτεμβρίου θα λάβει η χώρα η ακρόαση του κυρίου Χόγκαν από τις μισή ως τις μισή. Πρόκειται δηλαδή για τη δεύτερη ακρόαση ενός από αυτούς τους νέους επιτρόπους. Οπότε νομίζω πως υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θα ενδιαφερθούν και αναμένουμε ενδιαφέρον την ελογό ακρόαση. Επαναλαμβάνω λοιπόν τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 6.30 με 9 και μισή θα λάβει χώρα η ακρόαση του Επιτρόπου Φιλχόγκαν. Περνάμε ε, στο σημείο 6 της σας διάταξης, ε, ανταλλαγή δηλαδή απόψεων με την Eurofair και την European Aluminium, τις οργανώσεις δηλαδή από αυτούς τους ε, τομείς σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση στους τομείς του χάλιβα και του αλουμινίου. Η ανταλλαγή απόψεων με αυτές τις ενώσεις λαμβάνει η χώρα ανατακτά χρονικά διαστήματα σε σχέση με αυτό το θέμα, γιατί εδώ και πολύ καιρό ο εν λόγω κλάδος ε, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Ε, και μία από αυτές τις αιτίες, ε, από τις αιτίες για την κρίση, για τα προβλήματα, είναι ακριβώς η υπερπροσφορά χάλιβα στην παγκόσμια αγόργα. Και έχουμε και το παγκόσμιο βέβαια φόρουμ του χάλιβα, όπου συζητάτε ακριβώς η παγκόσμια μείωση της παραγωγικής ικανότητας χάλιβα χωρίς ωστόσο αυτό να, οδηγήσει, να έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στα επιθυμητά αποτελέσματα. Και από εκεί και μετά, από το 2018, έχουμε τις συμπληρωματικές ποσοστώσεις ε, από τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά το χάλιβα, που έχουν επιβληθεί δηλαδή στον, ε, στα δικά μας προϊόντα και αυτό βέβαια είχε επιπτώσεις στην αγορά χάλιβα στην Ευρώπη και από την ε, δική μας πλευρά εφαρμόσαμε αντίμετρα, αντισταθμιστικές ας το πούμε έτσι, ποσοστώσεις. προκειμένου να εξασφαλίσουμε κάποιες ε, προστασίες για τα προϊόντα μας που εξάγονται εκεί. Πράγμα που βέβαια και αυτό έχει τις επιπτώσεις του στις εξελίξεις ε, στην, στον κλάδο του χάλιβα και του αλουμινίου. Έχουμε τώρα κάποιες ε, διεθνείς δράσεις. Και ε, παρά τα όσα έχουν συζητηθεί σε σχέση με αυτούς τους δασμούς και τα αντίμετρα που έχουμε λάβει και εμείς δεν έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα ε, που να έχει οδηγήσει σε κάποια βελτίωση, ειδικότερα δηλαδή σε ό,τι αφορά το κλάδο του αλουμινίου, η παραγωγή μας είναι ακριβότερη ε, σε σύγκριση για παράδειγμα με την παραγωγή από την Κίνα. Άρα λοιπόν ο ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουμε από την Κίνα είναι πολύ σοβαρό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει και αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν λοιπόν μία σειρά από στοιχεία που συνθέτουν αυτή την προβληματική εικόνα του κλάδου του χάλιβα και του αλουμινίου στην Ευρώπη. Και προκειμένου λοιπόν να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα και προκειμένου να ακούσουμε και κάποιες ιδέες ως προς το τι μπορούμε να κάνουμε, έχουμε μαζί μας τον κύριο Καλντάτς ο οποίος είναι επικεφαλής ε, εμπορίου και εξωτερικών σχέσεων της Eurofair, ας σας βλέπω εκεί στο βάθος, και τον Τινόν Λάμπρετς, ε, ε, τον Διευθυντή Στατιστικών και Οικονομικών της, του Ευρωπαϊκού Κλάδου Αλουμινίου. Έχουμε επίσης τον κύριο Λεοπόλντο Ρουμπενάτσι από την Οργάνωση Άμυνας και Προστασίας του Εμπορίου και ο κύριος Κανάρντο επίσης ε, έχει προσκληθεί σήμερα εδώ που εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, την DigiTrade. Θα δώσω λοιπόν, θα δώσω καταρχήν τον λόγο στην Eurofair και στην European Aluminium. Thank you, Mr. Chair. Um, Ευχαριστούμε. Στο αλουμίνιο τώρα. Καλημέρα κυρίε και κύριοι και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σα ενημερώσω για την κατάσταση του κλάδου μας. Η, την αλουμινοβιοχανία στην Ευρώπη. Στον κλάδο μας υπάρχουν, εργάζονται περίπου 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι έμεσα και άμεσα με τζίρο 40 δις κάθε χρόνο. Υπάρχει αύξηση της ζήτησης αλουμινίου σε όλο τον κόσμο. Το χρειάζεται στο αυτοκίνητο, στο ποδήλατο, στο smartphone, στις ηλεκτρονικές συσκευές. Αυτές είναι λίγες από τις εφαρμογές τους οι τελικοί χρήστες, οι πιο σημαντικοί τελικοί χρήστες είναι η αυτοκιομηχανία, συσκευασία, πακέτα, πακέτα και, και πολλά καταναλωτικά προϊόντα. Είναι ανακυκλώσιμο προϊόν και ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάμπολες φορές με επανεπεξεργασία. Αυτό είναι πολύ καλό ε, εργαλείο για μια κυκλική οικονομία κατά συνέπεια. Η μετάβαση προς την, χαμηλ, οικονομία χαμηλού διοξιδίου του άνθρακα απαιτεί αλουμίνιο που μειώνει ε, τις δαπάνες σε διάφορους τομείς, ε, επιτρέποντας ευκολότερη κινητικότητα, καλύτερη αποδοτικότητα των συσκευασιών και μεγαλύτερη ε, εξοικονόμηση ενέργειας στα σπίτια. Το αλουμίνιο στην Ελλάδα είναι τρεις φορές ε, λιγότερο εντατικής χρήσης άνθρακα από το αλουμίνιο της Κίνας. Αυτό μας οδηγεί στον, ε, στη βασική απειλή του αλουμινίου στην Ευρώπη. Οι επιπτώσεις τη της υπερπαραγωγής της Κίνας που κάτι για το οποίο ε, σας προειδοποιούμε εδώ και χρόνια και που θέτει σε κίνδυνο την αγορά. η έκθεση του ΩΣΑ που δημοσιεύθηκε φέτος νωρίτερα τονίζει ότι η παραγωγή της Κίνας είναι ε, έχει ως αντίκτυπο ε, σε όλη την παγκόσμια αγορά με εκτιμήσεις που λένε ότι οι εξαγωγές από την Κίνα θα φτάσουν τα 60 δις ε, ανά τον κόσμο με διάφορες μορφές μείωσης της δαπάνης, φοροαπαλλαγές κλπ. Η παραγωγή αυξήθηκε από το 16% στο 57% μέσα σε δύο δεκαετίες. Αυτό οδήγησε σε τεράστια αύξηση της εξαγωγής των ή μη παρασκευασμένων προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, οι εισαγωγές από της Κίνας ε, φτάνουν στην αγορά σε χαμηλή τιμή, 30% περίπου λιγότερο από ό,τι τιμές αγοράς. Άρα, χτυπώντας παράνομα τον ανταγωνισμό των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αυτή η τάση που συνεχίζεται επιδίνωσε και, επι, και την κατάσταση και επιταχύνθηκε πρόσφατα. Λόγω του πολέμου μεταξύ, του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΙΠΑ και Κίνας, θύμα της οποίας μπορεί να είναι η Ευρώπη. Η, η επιρροή στους παραγωγείς είναι εμφανής. Κλείνουν διάφορες επιχειρήσεις από την Ευρώπη. Χωρίς ισχυρή δράση και άμεση δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των θέσεων εργασία στην Ευρώπη και μείωση της παραγωγής αλουμινίου στην Ευρώπη συνολικά. Πολλοί από του εταίρου της Ένωσης ήδη έχουν προχωρήσει περισσότερο από εμά στον τομέα αυτό, θέτοντα τι επιχειρήσει μα σε ακόμα μεγαλύτερη ε, αρνητική θέση. Αυτή τη στιγμή τα μέτρα για, τα, για τους τροχούς, ε, τους, ε, τα τα καλωδιφέρε και, τις μικρές, ε, και τους μικρούς ημάντες ε, ε, έχει σημαντική συνέπεια, κάτι που επηρεάζει πολλές μικιο, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δημιουργεί σοβαρά, σοβαρά οικονομικά ζητήματα. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του αθέμητου ανταγωνισμού χρησιμοποιώντας φερρυπίν νομικές δυνατότητες για την προστασία των προϊόντων της εν ώψη της ε, άμεσης απειλής. Επίσης πρέπει να λάβουμε δράση σε κάθε επίπεδο αντιμετωπίζοντας τις κρατικές ενισχύσεις, για παράδειγμα στην Κίνα. Ταυτόχρονα ζητούμε από την Ένωση να υποβάλει λύσεις σε περίπτωση που στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου δεν υπάρξει λύση. Ζητούμε εν ολίγης από την Ένωση να δείξει ότι είναι ικανή να προστατεύσει τη βιομηχανία της. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και ζητούμε την υποστήριξή σας στην προστασία και υπεράσπιση της αλουμινοβιομηχανίας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σαφή τα μηνύματα. Τι λέει η Κομισιόν για όλα αυτά. Λεοπόλτο. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για αυτές τις παρουσιάσεις. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεσλεύ για το μήνυμα ε, το οποίο μας περνάει σήμερα εδώ και το οποίο δεν ακούμε ε, συχνά, το ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει την απόφαση και είχε λάβει την απόφαση να παρέμβει στην καρδιά της κρίσης ε, στην αγορά του Χάλμπα. Νομίζω πως ε, έχουμε σημειώσει πολύ προσεκτικά τα όσα αναφέρθηκαν σήμερα εδώ ε, και θα ήθελα απλώς ε, να αναφέρω ένα-δυο στοιχεία τα οποία θεωρώ πολύ σημαντικά. Καταρχήν, το πρώτο σε ό,τι αφορά τι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε σε ό,τι αφορά το χάλυβα χάλιβα προέλευση εντονισίας. Από την 1η Οκτωβρίου ε, τα εν λόγω προϊόντα της Ινδονησίας θα καλύπτονται από τα προστατευτικά μέτρα σε ό,τι αφορά το χάλιβα. Και επίσης τον Αύγουστο ξεκινήσαμε μια έρευνα σε ό,τι αφορά το αντι dumping σε ό,τι αφορά τα προϊόντα αυτά προέλευσης και Ινδονησία αλλά και Κίνας. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό να σημειώσουμε εδώ ότι ότι η, Κίνα προσπαθεί ουσιαστικά με το δικό της τρόπο να δημιουργήσει αγορές σε τρίτες χώρες έτσι ώστε να αυξήσει την παραγωγή της και να μπορεί να εξάγει και περισσότερο και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει και εμείς να ε, δράσουμε αποφασιστικά και θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε ε, την συμβατότητα με τους κανόνες του Παγκόσμιου, Παγκόσμιου Οργανισμού ε, Εμπορίου από την πλευρά της Ινδονησίας. τώρα, σε ό,τι αφορά τα αντιμέτρα και τις ποσοστώσεις, από όσο γνωρίζω δεν, έχουν, δεν έχει σημειωθεί υπέρβαση μέχρι στιγμής. Μόνο για ένα-δύο προϊόντα έχει υπάρξει ε, υπέρβαση και για τους πρώτους δύο μήνες του 2019 τους συγκρίνουμε με τους δύο πρώτους μήνες του 2018 ε, όπου μπορούμε δηλαδή να κάνουμε μία ε, αντιπαραβολή των εισαγωγών, αλλά όχι σε ό,τι αφορά τα προστατευτικά μέτρα, τα αντίμετρα, βλέπουμε μείωση των εισαγωγών. Οπότε ε, τα όσα έχουμε κάνει εμείς πράγματι οδηγούν στα επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή την προστασία από τις εισαγωγές. Ωστόσο, από την ε, άλλη πλευρά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε στα προστατευτικά εμπορικά μέτρα ως επανάκια για τα ε, πάντα. Δηλαδή δεν μπορούμε για παράδειγμα σε ό,τι αφορά αθέμητες εισαγωγέ ή δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιου είδους μέτρα όταν υπάρχει μια μείωση γενικότερη της παγκόσμιας ζήτησης ή μια ύφεση ε, οικονομική. Άρα λοιπόν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά του χάλιβα είτε εξετάζονται αυτή την περίοδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε περιλαμβάνονται και στους πολιτικούς προσανατολισμούς ε, της ε, Προέδρου που έχει εκλεγεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε από τη δική μας πλευρά θα λάβουμε πολύ προσεπτικά υπόψη μας τα όσα αναφέρθηκαν. Τώρα έρχομαι στο αλουμίλιο. Ε, νομίζω πως εδώ θα πρέπει να εξετάσουμε από κοινού αυτό το ζήτημα. Δηλαδή ε, το, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ε, δεν έχουν κάποιο εμπόδιο στο να υποβάλουν τέτοιου είδου παράπονα σε ό,τι αφορά την προστασία του εμπορίου. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιου είδου προσφυγές που έχουν γίνει από την πλευρά μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ορισμένες φορές έχουμε καταφέρει ακριβώς να αντιμετωπίσουμε σε νομικό επίπεδο τέτοιου είδους πολιτικές στον χώρο του Χάλιβα και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε και το αντίστοιχο στο, στο αλουμίλιο. Αλλά για να το επιτύχουμε χρειαζόμαστε τα απαραίτητα δεδομένα, τα οποία δεδομένα μπορεί να μας παράσχει μόνο ο κλάδος του αλουμινίου. Οπότε θα πρέπει να ε, σκεφτούμε από γενού και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουμε είναι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε ε, αυτό που είπατε εσείς δηλαδή, τα μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μας, τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, στο μέγιστο δυνατό βαθμό και αυτό ακριβώς προτίθεται να κάνει η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Φρανσέσκο, τώρα έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως ε, ο κλάδος γνωρίζει πολύ καλά ότι βρισκόμαστε στο ε, πλευρό του ε, για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύο πολύ σοβαρές προκλήσεις που έχουν αναδειχθεί ε, και θα συνεχίσουν δυστυχώς να υπάρχουν. Δηλαδή η υπερβολική ικανότητα, παραγωγική ικανότητα της Κίνας και η πρόθεση από την πλευρά των ΗΠΑ να δημιουργήσουν καρτέλ ουσιαστικά σε ξένες αγορές. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στα όσα εμείς προσπαθούμε από την πλευρά της Digitrade να κάνουμε. Αυτό ήδη το ανέφεραν και οι συνάδελφοι από τον κλάδο του Χάλιβα. Δηλαδή ότι θα πρέπει να εξετάσουμε την πηχή των ε, πρώτων υλών ε, στην αλεξίδα τη παραγωγή αξία, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει που κάνουμε με την Ινδονησία για τη σύναψη μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Εδώ δηλαδή είμαστε πολύ προσεκτικοί, ούτω ώστε να διασφαλίσουμε ότι η πρόσβαση στι πρώτε ύλε, όπω το Νικέλιο για παράδειγμα, που είναι εξαιρετικά σημαντικέ για τον τομέα του αλουμίνου, ε, είναι διαθέσιμες και θα έχουμε πρόσβαση σε αυτές μέσα σε αυτή τη νέα συμφωνία. Τώρα, σας αναφέρω όλα αυτά και βέβαια μπορείτε να μας πείτε και εσείς και να μας ρωτήσετε πώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις, αλλά από εκεί και μετά θα πρέπει να πούμε ότι είναι θεμελιώδης σημασίας ε, αυτό που το γεγονό ότι δηλαδή θα πρέπει να λάβουμε από τώρα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε μελλοντικέ προκλήσει. Καταρχήν θέλουμε ε, καλύτερη επιβολή τη νομοθεσία και γι' αυτό η ε, νέα πρόεδρο Βαντρελάιν έχει αποφασίσει ότι θα υπάρξει ένα ειδικό αξιωματούχο σε ό,τι αφορά ακριβώ την επιβολή τη νομοθεσία. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζουμε λοιπόν την προστασία των δικαιωμάτων. Ε, δεύτερο σημείο τώρα. Γνωρίζουμε πω το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα δεν επαρκεί. Και γι' αυτό έχουμε ήδη ξεκινήσει την αναδιαπραγμάτευση αυτών των κανόνων έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαπραγμάτευσή του στον, στον, στον ΠΟΕΜ. Και έχουμε ξεκινήσει και μια διαπραγμάτευση με του αδέλφου από τι ΗΠΑ και την Ιαπωνία, προκειμένου οι νέοι αυτοί κανόνε να μπορέσουν να καλύψουν όλα τα προβλήματα στρέβλωση του εμπορίου που δημιουργούνται ακριβώ από την υπερβολική παραγωγική ικανότητα τη Κίνα. Ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η χάραξη τη σωστή πολιτική ξεκινάει από εμά, από εδώ. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμεί έχουμε ξεκινήσει μια εξέταση ε, του πώς μπορούμε να δούμε το, πώς ασκούνται ε, οι διάφοροι μοχλήπες σε ό,τι αφορά την εσωτερική μας αγορά, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν από την υπερβολική παραγωγική ικανότητα. Όλα λοιπόν αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη μας, αλλά επιτρέψτε μου να τονίσω δύο πτυχές. Πρώτον, η εμπορική πολιτική είναι πολύ σημαντική, αλλά δεν είναι ε, με απανάκια. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί να μας επιτρέψει να, να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα. Και γι' αυτό η πρόεδρο Βαντερ έχει τονίσει εδώ δύο πολύ σημαντικές επιτυχίες. Η μία είναι το ότι θα πρέπει να αξιοποιούμε όλα τα εργαλεία τη εμπορική πολιτική που έχουμε έτσι ώστε να προστατεύσουμε αυτού του δύο πολύ σημαντικού βιομηχανικού κλάδου και ταυτόχρονα θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μα την περιβαλλοντική πτυχή σε ό,τι αφορά δηλαδή ε, και του ε, φόρου ε, άνθρακα, πομπών Άρα λοιπόν θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλε τι δυνατότητε που έχουμε στη διάθεσή μα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι δύο προκλήσει οι οποίε θα συνεχίσουν να υφίστανται και στο εγγυσμένο. Και, θα... και είμαστε διατεθειμένοι από τη δική μα πλευρά να συνεργαστούμε και με του Αμερικανού φίλου μα. Έχετε δει ε, πόσο ξεκάθαρη ήταν η δική μας ε, απάντηση σε δύο-τρία ε, μέτρα που λύθησαν και είδατε και το τι χρειάστηκε να κάνει και ο πρόεδρος ε, Γιούνκερ ε, σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ έτσι ώστε για παράδειγμα να αποφύγουμε την επιβολή τέτοιου είδου μέτρων σε ό,τι αφορά την αυτοκίνητο βιομηχανία. Και αυτή λοιπόν η κατηγορηματική στάση την οποία έχουμε οθετήσει ε, νομίζω πως θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. θα ολοκληρώσω τώρα με ένα σχόλιο. παρόλα αυτά τα νέα διπλωματικά εργαλεία που είχαμε στη διάθεσή μα για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη ε, μεγάλη παραγωγική ικανότητα, ε, ταυτόχρονα είχαμε και την ε, υποστήριξη από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί κάθε φορά που κάνατε επισκέψει στην Κίνα, ε, ασκήσατε πιέσει, οι οποίε πραγματικά μα βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό. Παρότι δηλαδή αυτή η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην Κίνα συνεχίζει να υφίσταται. Ήδη τα όσα έχετε κάνει έχουν επιφέρει αποτελέσματα, οπότε θα ήθελα να σας καλέσω να συνεχίσετε τις προσπάθειές σας ε, όπως σας ανέφερα τώρα και εκπρόσωποι από τους δύο ε, κλάδους, να συνεχίσετε λοιπόν αλλά και να μας ε, παράσχετε και περαιτέρω εργαλεία και περαιτέρω μοχλούς άσκησης πιέσεων έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την, ε, την δημιουργία καρτέλα από την πλευρά των λοιπόν σε ξένες αγορές και την υπερβολική παραγωγική ικανότητα της Κίνας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 Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ και τους δύο εκπροσώπους των κλάδων και την Επιτροπή για την ενημέρωση. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητούμε το θέμα αυτό και τις προκλήσεις που σχετίζονται με αυτό. Θέλω να τονίσω ωστόσο ένα πρόβλημα που δεν έχουμε συζητήσει ουσιαστικά. Πώς οι βιομηχανικές πολιτικές στις χώρες που επηρεάζονται ασχολούνται με την παραγωγή χάλιβα στην ουσία. Αν δείτε στην Κίνα χτίζουν νέες πόλεις παντού και είναι σαφές ότι χρειάζονται χάλιβα. Θα μπορούσε η Ένωση να καλύψει τις ανάγκες αυτές της Κίνας. Δηλαδή πρέπει να λάβουμε υπόψη τις εθνικές στρατηγικές της Βραζιλίας, της Κίνας, των ευρωπαϊκών χωρών, των ΗΠΑ και πώς αντιμετωπίζουν στρατηγικά την αύξηση, τη μείωση της ζήτησης. Αν δείτε τα νούμερα για το χάλιβα, οι εισαγωγές από την Ένωση τα τελευταία χρόνια είναι σαφές ότι μειώθηκαν. Σχετίζονται ωστόσο με τη γενικότερη κατάσταση βασικές εισαγωγές της Ένωσης προέρχονται από την Τουρκία, που αντιδρά στην ε, αύξηση των ε, δασμών από τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, για την ευρωπαϊκή αγορά. Μετά έχουμε τη Ρωσία, την Ουκρανία, Κίνα 7%, Νότιος Κορέα 6%, Βραζιλία 6%, Ινδία 6%. Η εικόνα που έχουμε δίνει μια διαφορετική συνολική εντύπωση. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε το πρόβλημα σε πιο μάικρο επίπεδο και με βάση τις ανάγκες και με βάση τις εθνικές στρατηγικές και με βάση τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Συνάδελφοι, πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο. Δύο λεπτά παρακαλώ να τα σέβεστε. Σούστε. Σα ευχαριστώ και ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του εκπροσώπου ε, των ε, κλάδων. Δύο ε, στοιχεία θα ήθελα εγώ να αναφέρω από την πλευρά μου. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τα προστατευτικά μέτρα, τα οποία λήφθησαν σε συνέχεια των δασμών που επέβαλαν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, πρόσφατα έγινε μια εξέταση αυτών των μέτρων και αυξήθηκαν οι ποσοστώσει. Μα αφού λέμε ότι δεν εξαντλήθηκαν στο ε, πλήρωση αυτέ οι ποσοστώσει, και αφού βρισκόμαστε ε, στα πρόθυρα μιας οικονομικής ύφεσης, γιατί αυξάνουμε αυτές τις ποσοστώσεις οι οποίε ουσιαστικά δημιουργούν ακόμα περισσότερε επιέσει στην αγορά. Και αυτό που είπε ο συνάδελφο Σόλη είναι πολύ σημαντικό, ότι δηλαδή ε, ακριβώ ε, η, η ουσιαστικά οι παρεκτροπέ οι οποίε λαμβάνουν χώρα στο εμπόριο είναι εκείνε που δημιουργούν το πρόβλημα. Δηλαδή, όχι ακριβώ η αλλά ακριβώ αυτό που συμβαίνει μέσω τη Τουρκία. Από εκεί και μετά, εκείνο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα, ειδικότερα και μετά από τι διαδηλώσει του Σαββατοκύριακου, τι θα συμβεί σε επίπεδο του Green Border Adjustment, γιατί έχουμε ε, και όλες αυτές τις διαρροές, ε, αν θα αυτό το carbon leakage, λόγω ακριβώς και των ε, τιμών στους δικούς μας κλάδους οι οποίες έχουν αυξηθεί ακριβώς λόγω του συστήματος εμπορίας εκπομπών που έχουμε επιβάλει και όπου θα πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη αποζημίωση ακριβώς για να αντισταθμίσουμε ε, τις ε, ε, τιμές στις αγορές εκείνες όπου δεν επιβάλλεται ένας τέτοιος φόρος από διοξιδίου του άνθρακα. Άρα λοιπόν αυτά που είπε και ο κ. Αμπουδικόφα ότι δηλαδή θα πρέπει να γίνει μια εξέταση κατά πόσο τα εν λόγω μέτρα είναι συμβατά με, τις, με τους κανόνες του ΠΟΕ είναι κάτι που θα πρέπει να το εξετάσουμε περαιτέρω και να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες για τις δύο κλάδους. Πρόεδρο, ε, τώρα έχουμε ένα πρόβλημα γιατί υπάρχουν 10 ακόμα συνάδελφοι που έχουν ε, ζητήσει το λόγο, πράγμα το οποίο θα σήμαινε 20 ακόμα λεπτά για τη συζήτηση. Α, όχι, 9 τώρα. 1,5 λεπτό ο, ο καθένα θα έχει το λόγο, ο κ. Μορέλ.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 Κατάινεν. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ τους ομιλητές για την παρουσίαση των θεμάτων στον τομέα. Είναι σαφές ότι οι εξελίξεις είναι σημαντικές και πρέπει η Επιτροπή να αντιδράσει στις διακυμάνσεις των τιμών στην παγκόσμια αγορά με τους δασμούς, για παράδειγμα. Αυτό σχετίζεται και με την ε, παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα στην ε, Ινδονησία για παράδειγμα η παρουσία του διοξιδίου του άνθρακα είναι πολύ σημαντικότερη από ό,τι στην Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω για το πώς ε, περισσότερο για αυτό το κείμενο για την φορολογία του διοξιδίου του άνθρακα που περιέλαβε η κυρία Φοντελάιν στο πρόγραμμα των 100 ημερών, των 100 ημερών της. Πού πηγαίνουμε σε αυτό. Καλημέρα, λέει η κυρία Αγγιλάρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την ΕΡΟΦΕΡ που ήρθε εδώ για να μας ενημερώσει για την παρούσα κατάσταση στο, στο, στους δύο κλάδους αυτού στην Ένωση και να ευχαριστήσω την Γραμματεία και τα μέλη που έρχονται εδώ ξανά για να τονίσω τα μέτρα που είχαμε ήδη συζητήσει για τα μέτρα προστασίας της ευρωπαϊκής αγοράς και τις στρεβλώσεις που, που είχαν προκύψει στο παρελθόν από τις εισαγωγές από Κίνα. Ω εκπρόσωπο τη Ισπανία εδώ θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που συνιστά για μα αυτά τα μέτρα διασφάλισης που μειώνουν μια σοβαρή απειλή για ένα σημαντικό κλάδο για την οικονομία και την απασχόληση στη χώρα μου. Η σημασία αυτή είναι μεγάλη όχι μόνο για την Ισπανία αλλά και για άλλες χώρες. Γερμανία, Ρουμανία, Τσεχία, Ελλάδα, πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κλάδος είναι θεμελιώδης για μας και θέλω να υποστηρίξω απόλυτα τέτοιες αποφάσεις όπως και αυτήν για την μετατροπή των προσωρινών σε οριστικά μέτρα. Είναι σημαντικό να μην υπάρξουν αδικαιολόγητες αυξήσεις εισαγωγών, οι συνέπειες των οποίων στην ευρωπαϊκή οικονομία θα ήταν εξαιρετικά στρεβλές. Ω μέλο της ομάδας των ε, συντηρητικών και εκπροσωπώντα το Vox, το κόμμα Vox, η εντολή που έλαβα από τους πολίτε της Ισπανίας είναι να προστατεύσω το διεθνές εμπόριο χωρίς όμως να θέσω σε δυσμενέστερη φάση την ευρωπαϊκή μορφή παραγωγής, κάτι που συμφωνούμε, επί το οποίο συμφωνούμε όλοι. Δεν θα υποστηρίξω μέτρα τα συν, οι συνέπειες ε, και επιπτώσεις των οποίων θα πλήττουν ε, την απασχόληση και την οικονομία της χώρας. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ με... Μου άρεσε πολύ όταν αναφέρθηκε από την Επιτροπή ότι η κυρία Βοντελάιεν θέλει να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα πολιτικών ε, ε, για την ευρωπαϊκή παραγωγή. Μπορεί να μας πούν λίγα περισσότερα πράγματα. Τι κίνητρα μπορεί να τεθούν από την άποψη της Επιτροπής ούτως ώστε ο κλάδος να βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα ε, της παραγωγής χάλιβα. Είδαμε προοδευτικά παραδείγματα στον κλάδο του αλουμινίου κυρίως στην παρουσίαση που έγινε. Γνωρίζω ωστόσο ότι και στις σκανδιναβικές χώρες η παραγωγή χάλιβα γίνεται όλο και πιο ενεργοαποδοτική. Θέλω λοιπόν να ακούσω λίγο περισσότερα πράγματα από τον κλάδο. Τι μπορούμε να πετύχουμε την επόμενη πενταετία στον τομέα αυτό. Γιατί προφανώς μακροπρόθεσμα αυτό θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Αν δεχθούμε, όπως το δέχομαι εγώ, ότι θα θελήσει η Ένωση να έχει ισχυρότερη δράση έναντι αυτών που υστερούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Κάνας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι προφανές ότι ο κλάδος ε, του Χάλιβα και του αλουμινίου είναι στρατηγική σημασίας για την Ένωση. Ταυτόχρονα είναι κλάδοι που απαιτούν εργατικό δυναμικό ποιότητας που πρέπει να προστατεύσουμε. Μιλήσαμε για εμπορικές ροές, για υπερπαραγωγή, για dumping, αλλά λίγο είδαμε πώς όλα αυτά επηρεάζουν την απασχόληση, που είναι θεμελιώδους σημασίας στην ουσία. Εγώ είμαι εδώ για να συζητήσω και συνέπειες που στρατηγικές όπως αυτή της Κίνας ή των ΗΠΑ ε, αποσκοπούν όχι ε, στην, ε, στο να πλημμυρίσουν τον κόσμο με δικό τους χάλιβα, που είναι μια στρατηγική, δεν είναι τακτική μόνο. Τι συνέπειες έχει τελικά η, η αργή ή η ανεπαρκής απάντηση της Ευρώπης στις εισαγωγέ για την απασχόληση. Είναι μια πολιτική στάση, διότι ε, υπήρξε έλλειψη αποτελεσματικής αντίδρασης εκ των ε, προτέρων. Ρωτώ λοιπόν, έχετε σκεφτεί την ταχύτητα λήψης μέτρων που προστατεύουν την ευρωπαϊκή οικονομία, επίσης όμως και τον κλάδο, όταν δεν εκμεταλλεύεται την κατάσταση αυτή για να επενδύσει, για να δει πώς μπορεί να αντιδράσει ο κλάδος όταν οι κάποιοι αντιδρούν ταχύτατα και ε, α, αμέσως ενώ άλλοι καθυστερούν χωρίς να επενδύουν. Ευχαριστώ. Γιάννη Μαρή. Ευχαριστώ πρόεδρε για την ενημέρωση. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με το ρόλο του νέου ε, επικεφαλής ε, της επιβολής του νόμου που ανήγγειλε η κυρία Βαντελάιεν. Πώς ε, βλέπετε να είναι αποτελεσματικός ο ρόλος αυτός και συμπληρωματικός σε αυτόν που έχουν οι διεθνείς δομές Φερπίνο ΠΟΕ. Δεύτερον, η Επιτροπή περιμένει ότι αυτό θα έχει, θα οδηγήσει στην αναγκαία αύξηση του προσωπικού για να είναι αποτελεσματική η δράση αυτού του ρόλου. Σαλίνη. Δύο συγκεκριμένα ερωτήματα θα ήθελα να θέσω. Ε, σε ό,τι αφορά την ε, απομένουσα ποσόστοση ε, και σε ό,τι αφορά τη στοχευμένη προσέγγιση, τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε σε ό,τι αφορά αυτή την ποσόστοση που παραμένει και μετά. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιε είναι οι επιπτώσει του Brexit σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα προστατευτικά μέτρα που έχουμε λάβει. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μπέντ. Μια συγκεκριμένη ερώτηση προς την Επιτροπή. Το border adjustment είναι προφανώς κάτι δύσκολο να υλοποιηθεί. Γιατί εδώ πρέπει να έχουμε ένα tax carbon που δύσκολα θα μπορέσει να υλοποιηθεί γιατί θα απαιτήσει ομοφωνία στο Συμβούλιο. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι η Επιτροπή κρίνει πως είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στις ε, μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες μια υποχρέωση του αντισυμβαλόμενου να έχει ένα σύστημα cap and trade αντίστοιχο με το δικό μας. Θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι μια μείζον ε, εξέλιξη αυτή. Την ίδια ερώτηση τη θέτω και στους εκπροσώπους του κλάδου. Θα μπορούσε μια τέτοια λύση να λύσει κάπως το πρόβλημα. Τελευταία, τελευταία ερώτηση, ο κύριος Μπορά. Ναι, ευχαριστώ πολύ σύντομα. Τρία σύντομα ερωτήματα θα θέσω. Καταρχήν, μέτρα την dumping. Από ό,τι βλέπουμε, ουσιαστικά η Τουρκία εμ, καταφέρνει να τα προσπεράσει, α το πούμε έτσι, και η Ινδονησία το ίδιο. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το καταπολεμήσουμε αυτό. Μετά, σε ό,τι αφορά τα προστατευτικά μέτρα των ΗΠΑ προκειμένου υποτίθεται να προστατεύσει τα συμφέροντά τη αυτή η χώρα. Τι μπορούμε να κάνουμε τόσο ώστε να αντιδράσουμε απέναντι στι ΗΠΑ, πώ μπορούμε δηλαδή να πιέσουμε την Αμερικανική πλευρά να διαπραγματευτεί μαζί μα. Ε, και από εκεί και μετά αυτό το Carbon Adjustment Tax, ε, αυτό ο φόρο δηλαδή για την προσαρμογή σε ό,τι αφορά τι εκπομπέ του άνθρακα, πώ συμβιβάζεται με του κανόνε ε, του ΠΟΕ. Πρόεδρο, δεν ξέρω κατά πόσο θα λάβετε κάποια απάντηση στην τελευταία σα ερώτηση, αλλά για να δούμε. Λοιπόν, θα δώσω τώρα το λόγο στους εμπειρογνώμονες τρία λεπτά. Πάνω κάτω. Αλλά βέβαια τα περισσότερα ερωτήματα τέθηκαν ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο εκπρόσωπος της Eurofair έχει πρώτος ε, το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ. Ε, θα απαντήσω κάποια ερωτήματα στα οποία μπορώ να απαντήσω. Καταρχήν, κύριε Σόλτσε, να σας πω, για να διορθώσω κάτι που είπατε, είπατε ότι υπάρχει κατά τα τελευταία χρόνια μείωση των εισαγωγών στο χάλιβα. Το αντίθετο συμβαίνει με βαστατεστικά στοιχεία. Αυτό που συμβαίνει είναι πως η πηγή των εισαγωγών έχει ε, αλλάξει. Δηλαδή, η Κίνα έχει ε, μειώσει τις εξαγωγές της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτή η μείωση έχει ε, ουσιαστικά τη σταθμεί και με το παραπάνω από άλλες χώρες οι οποίες έχουν υπερπαραγωγή σε σχέση με τις ανάγκες της εσωτερικής τους αγοράς. Και ο λόγο χώρες αυτές είναι η Τουρκία. Γνωρίζουμε εκεί τις αγορές ε, που υπάρχουν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ε, η Ρωσία, λοιπόν και από εκεί και μετά και η Κίνα για κάποια προϊόντα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο του υπάρξουν λήψεις ε, χάλιβα στην ευρωπαϊκή αγορά. Ε, αντιλαμβανόμαστε ότι ορισμένοι εισαγωγεί έχουν πει ότι ακριβώ με την εφαρμογή αυτών των προστατευτικών μέτρων θα μπορούσε να προκύψει έλλειψη στην προσφορά χάλιβα. Ε, ε, ε με βάση και το έγγραφο κοινοποίηση στον ΠΟΕ έχει εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο, αλλά έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά στοιχεία που να το υποστηρίζουν. Ε, η δική μας εμπειρία είναι ότι συχνά ακούμε τέτοιου είδους επιχειρήματα, αλλά ουσιαστικά εδώ ε, βασίζονται σε μια σύγχυση ανάμεσα στο να υπάρχει τέτοια πραγματική έλλειψη αφενός και από την άλλη το να έχουμε ουσιαστικά την φτηνότερη παραγωγή χάλιβα. Ε, από όσο έχει υπάρξει ε, ποτέ. Μετά, ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της πολιτικής μας ουσιαστικά, πραγματικά το χαιρετίζουμε γιατί βλέπουμε να υπάρχει μια διαφορετική νοοτροπία. Γιατί μέχρι στιγμής η εμπορική πολιτική βασιζόταν στις υφιστάμενες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, FTA δηλαδή. Ε, οι συμφωνίε όμω οι οποίε ουσιαστικά υπονομεύουν την πειθαρχία, αν θέλετε, που ε, επιβάλλουν οι κανόνε του ΠΟΕ. Βέβαια, θα πρέπει να υπάρξουν τώρα νέοι κανόνε, οι οποίοι ακριβώ θα χρησιμοποιούνται και θα είναι δυνατόν να υποστηρίζονται από όσου καλύπτονται από αυτού του κανόνε. Αλλά δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τις συμφωνίες αυτές και ε, το κατά πόσο τελικά οι κανόνε του εφαρμόζονται στην πράξη αλλά έχουμε να κάνουμε και με τον ίδιο τον ε, Όπως αναφέραμε στο παράδειγμά μας δηλαδή, με, τις εξαγωγικές, ε, με τους εξαγωγικούς περιορισμούς της ε, Ινδονησίας, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούν να εφαρμοστούν και λαμβάνοντας υπόψη το τι συμβαίνει στον κλάδο μας θα πρέπει να εφαρμοστούν. Ευχαριστούμε. Τώρα, λέει ο πρόεδρος, τώρα ο εκπρόσωπος από τον κλάδο αλουμινίου. Σε ό,τι αφορά ε, την ένταση ενέργειας ε, ε, σε αυτό το τομέα, ναι, γνωρίζετε πως το είναι ενεργοβόρος ο κλάδος μας, δηλαδή το 40% του κόστους για την παραγωγή αλουμινίου είναι ενεργειακό, οπότε σε κάθε περίπτωση θέλουμε να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας και με το carbon leakage λοιπόν έχουμε χάσει ακριβώς αυτό το 1 τρίτο Οπότε κατά συνέπεια θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε καλύτερες επενδύσεις όπως για παράδειγμα αυτό το project με την ε, μπαταρία αλουμινίου αφού εκεί θα ε, η θήκη στην οποία θα βρίσκεται μέσα η μπαταρία θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο. Άρα λοιπόν κάνουμε ό,τι μπορούμε από την πλευρά του κλάδου για να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργεια μα. Επίση, συμφωνούμε με αυτό που υπόθηκε ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή εμπορική πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα νομικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται τα μέτρα για την καταπολέμηση των κρατικών ενισχύσεων. Γιατί τέτοιου είδου ενισχύσει, για παράδειγμα στην κοινωνική νοσοποίηση, οι οδηγούν ε, στην υπερβολική παραγωγική ικανότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτόν τον αξιωματούχο, ο οποίο θα οριστεί για την επιβολή τη νομοθεσία, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώ θα κάνει, αλλά ενδεχομένω θα μπορούσε να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο ακριβώ του κανονιστικού πλαίσιου του ΠΟΕ. Δεν ξέρω αν απάντησα με αυτόν τον τρόπο στα ερωτήματα που τέθηκαν αλλά πραγματικά πρόκειται για ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα. Ευχαριστώ. Αν υπάρξουν συμπληρωματικές ερωτήσεις μπορείτε να απαντήσετε. Δεν είναι εύκολη δουλειά να απαντήσει σε όλα αυτά η Επιτροπή. Υπήρχε έτοιμα για δράση. Λοπόλτο. Ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τις κυρίες και τους κυρίους βουλευτές για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έγινε. Σημειώσαμε πολλά πράγματα και έχουμε και πολλά να σκεφτούμε. Πρώτα πρώτα, για όλες αυτές τις συζητήσεις για το φόρο border adjustment, την ε, επιβάνηση άνθρακα κλπ. Αφήστε μας να δουλέψουμε, να σκεφτούμε, να εξετάσουμε τις διάφορες εναλλακτικέ. Μεταξύ αυτών την κεντρική ερώτηση είναι σύμβατα με τον μπορεί όχι τα μέτρα αυτά, ούτω ώστε να... και μόλις έχουμε κάτι που θα μπορούμε να το παρουσιάσουμε, θα το παρουσιάσουμε και ενώπιόν σας. Αλλά θέλουμε να το σκεφτούμε προσεκτικά. Τώρα, μέτρα προστασία, μέτρα διασφάλισης. Αυξήσαμε το επίπεδο ποσοστώσεων δασμών γιατί είναι υποχρέωση μέσω του ΠΟΕ. Η διασφάλιση είναι προσωρινό μέτρο που πρέπει να συνοδεύεται από ένα στοιχείο προοδευτικής απελευθέρωσης. Το πρόβλημα δεν είναι κατά την απόψή μας ε, τα ποσοστά δασμών, αλλά ότι κάποιες χώρες έχουν καταχραστεί του συστήματος και γι' αυτό κατά την άποψή μας ε, έχουμε εξετάσει διάφορα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα επιτρέπεται πλέον η κατάχρηση του συστήματος μεταξύ αυτών και το θέμα της διαχείρισης των ποσοστώσεων και των υπολοιματικών ποσοστώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Χρειαζόμαστε περισσότερους κανόνες, αυτό είναι σαφές. Όχι αναγκαστικά στη φάση αυτή εξετάζοντας και την ε, εσωτερική νομοθεσία για τα DDI και σε πολυμερές επίπεδο. Χρειαζόμαστε αυστηρότερους κανόνες για τις ενισχύσεις και χρειαζόμαστε τους κανόνες αυτές σε παγκόσμιο επίπεδο, πολυμερός δηλαδή. Και αυτό είναι μια ισχυρή δέσμευση που έχουμε και με τη ΣΥΠΑ και με την Ιαπωνία, αλλά και με την Κίνα. Το θέμα της έλλειψης ε, χάλιβα είναι σημαντικό ζήτημα. Μιλούμε τώρα με τον κλάδο παραγωγής αλουμινίου και χάλιβα. Αλλά ξέρετε ότι υπάρχει και μια μεγάλη βιομηχανία χρηστών στην που δεν θέλει αύξηση των τιμών πολύ. Το εγχείρημα λοιπόν, αν είναι, το, η συζήτηση αν είναι μέτρο αντι-dumping ή μέτρο αντι-subsidy, είναι ε, να σεβαστούμε τα, τις ισορροπίες παγκόσμιας οικονομίας, άρα και τα συμφέροντα των τελικών χρηστών. Εν τέλει, το θέμα του chief enforcer, του βασικού επιβάλλοντος ε, την νομοθεσία. Είναι προφανές ότι η προσωπικότητα αυτή θα πρέπει να μπορεί να δράσει. Άρα το άτομο αυτό να έχει επαρκείς πόρους για να ασκεί τα καθήκοντά του ή της. Ευχαριστώ. Φρανσίσκο. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μπούτιχόφερ. Χρειαζόμαστε εργαλεία, μοχλούς για να συζητούμε με την Κίνα. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα με ακούσετε να λέω ότι οι πρωτοβουλίες όπως ένα μέσο διεθνών, διεθνών προμηθειών θα μπορούσε να παράσχει αυτό το χώρο διαπραγματεύσεων που χρειαζόμαστε με την Κίνα. Στον κύριο Σόλτς, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν ανάγκες ανάπτυξης των εταίρων μας. Το πρόβλημα με την Κίνα είναι ότι η Κίνα έχει αυξήσει και το δυναμικό της πολύ περισσότερο από τις ανάγκες ανάπτυξη της κατά 500 εκατομμύρια τόνους από το 2000 που είναι ακριβώς η, η υπερπαραγωγή αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς τούτο έγινε όχι ακολουθώντας τις απαιτήσεις της αγοράς αλλά τις την καθοδήγηση του κράτους που δημιούργησε ένα σοβαρό πρόβλημα που το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι Κινέζοι. Και το πρόβλημα είναι ότι παρότι στη φάση αυτή η δυναμικότητα της κινέζικης αγοράς είναι μεγάλη, δηλαδή χρησιμοποιούν πολύ παραγωγή οι Κινέζοι. Όταν πέσει η αγορά που είναι κυκλική, θα έχει μια μεταφυσική πραγματικότητα. Τι θα κάνει αυτή η παραγωγή, πού θα πάει. Το είδαμε και στο παρελθόν. Θα ξεχυθεί στην υπόλοιπη παγκόσμια αγορά. Και αυτό είναι ένα, μια βασική απειλή για την επιβίωση του ευρωπαϊκού κλάδου. Όχι γιατί δεν είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά γιατί οι εξαγωγές θα πρέπει να γίνουν, θα γίνουν μάλλον σε αθέμητες ε, τιμές. Συμφωνώ και με τον κύριο Σόστ για το Global Forum. Είναι ένας σημαντικός δρόμος για να συζητήσουμε την αύξηση, την υπερπαραγωγή. Η Υπουργική Σύνοδος που θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου θα έχει καθοριστικό ρόλο. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε για την επέκταση αυτού του φόρουμ και την διατήρηση ενός ισχυρού φόρουμ που θα μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και μπορώ να σας πω το εξής. Εκεί θα δείξουν όλοι τα χαρτιά τους οι Κινέζοι συνάδελφοι που ε, ε, περνούν αρνητικά μηνύματα ακόμα και στη σύνοδο της Οζάκα για την επέκταση του φόρου θα δείξουν, θα πρέπει να δείξουν αν είναι υπέρ, πραγματικά υπέρ ή όχι της πολυμερούς συνεργασίας. Αν θέλουν να τελειώσουν το φόρο θα το δείξουν. Ή θα πρέπει να δείξουν ότι όντως ενδιαφέρονται για να παίζουν με τους κανόνες. Άρα, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα που είναι αβέβαιο, θα πρέπει να ε, δούμε τις συνέπειες. Ότι δηλαδή όταν μιλάμε για πολυμερή συνεργασία πρέπει να δείξουμε και την ε, υποστήριξή μας. Ένα σχόλιο επίσης. να πω στον κύριο Ριτζιμέντη και στον κύριο Ντάντε, δεν είναι, μόνοι, δεν είναι μόνος του ο κλάδος. Εμείς συνεργαζόμαστε στενά για να λύσουμε όλα τα προβλήματα όπως μπορούμε. Προφανώς υπάρχουν ρυθμίσεις, ισχυρές, δυνατές ρυθμίσεις προστασία του περιβάλλοντο στι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταλάβουμε υπόψη για τι διαστάσει του κύριου Χάνσεν. Και εγώ μία ερώτηση για το μέσο IPI. Όλοι λένε ότι είναι χρήσιμο. Όπως ξέρετε η Επιτροπή ήταν ενεργή, δραστήρια, και ο Σκασπάρη Κασπάρη θεωρούσε ότι έτσι μπορεί να ξεπεραστεί το μπλοκάρισμα στο Συμβούλιο. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για το τι γίνεται στο Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Η εντύπωση που έχω είναι ότι το Συμβούλιο στη φάση αυτή κινείται και υπάρχει μία πιθανότητα να προχωρήσει στην υιοθέτηση της νομοθεσίας.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 Η τρίτη περιφέρεια που έχουμε, όπου δεν έχουμε επάλα, δύο χώρες που εφαρμόζουν την EPA, Ακτήλεφαντοστού και Γκάνα, σε διμερές επίπεδο, γιατί με την περιφέρεια αυτή οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν και αυτές το 2014. Μία χώρα, η Νιγηρία, δεν έχει υπογράψει την Περιφερειακή Συμφωνία συζητούμε ακόμα μαζί του, αλλά είναι ασαφέ κατά πόσον θα, το θα την υπογράψουν ή όχι. Ταυτόχρονα αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε την συμφωνία με τι άλλε δύο χώρε. Ακτή ελεφαντό του Γκάνα δεν ήταν επιλέξιμε πλέον για ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά τη Ένωση. Είχαν γίνει χώρε μέση οικονομία. Δημιουργήσαμε λοιπόν την EPA μαζί τους εδώ και τρία χρόνια. Η τελευταία χώρα με την οποία έχουμε μία διαπραγμάτευση είναι το Καμερούν στη Δυτική Αφρική, η μόνη χώρα με την οποία, που είναι και σημαντικός παίκτη για μας. 14 χώρες συνολικά που όπως είπα έχουν πρόσφατη εφαρμογή, 2-3 χρόνια κατά βάση υλοποίηση, άρα είμαστε στο ξεκίνημα ακόμα για να δούμε κατά πόσον η συμφωνία δουλεύει ή όχι. Αν δείτε όμως τα εμπορικά στοιχεία, κοιτάμε τα στοιχεία του 18 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, στις 14 χώρες EPA η αύξηση των εξαγωγών ήταν 5 με 6%. Διαφέρει αυτό από χώρα σε χώρα. Συνολικά όμως η τάση είναι ανωδική. Δύο λόγια τώρα για την ε, μετά κοτονού κατάσταση. Το συνολικό πλαίσιο είναι μια συμφωνία συνολικού πλαισίου με τις χώρες ΑΚΕ. Δεν είναι εμπορική συμφωνία. Καλύπτει πολύ περισσότερους τομείς από το εμπόριο, αλλά μας παρέχει σημαντικά στοιχεία. Κατά βάση τα ουσιαστικά ε, στοιχεία που χρειαζόμαστε και σε άλλες συμφωνίες. Η διαπραγμάτευση λοιπόν για μας είναι σημαντική. Επίσης παρέχει μεγαλύτερη συνεργασία με όλες αυτές τις χώρες, ιδίως τις χώρες που δεν έχουν μία EPA μαζί μας. Θέλουμε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για την κατάσταση μετά το Κοτονού. Καλά πάνε. Άλλοι βέβαια ασχολούνται με τη διαπραγμάτευση κατά βάση, η DEVCO, αλλά έχουμε κάποια κοινά στοιχεία. Είναι ένα κεφάλαιο και τρεις πυλώνες αναπεριφέρεια. Εμείς Το παρακολουθούμε στενά. Τελευταίο θέμα, σημαντικό για το Κοινοβούλιο νομίζω και για μας ως Επιτροπή, ο ρόλο τη κοινωνία των πολιτών. Εδώ ασκούμε πίεση στου εταίρου στη συμφωνία EPA. Οι διαπραγματεύσει, βέβαια, οι συμφωνίε ε, ήταν διαφορετικά, είχαν διαφορετικά χρονικά ορόσημα. Σε κάποιε υπήρχε εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, μεγαλύτερη ή μικρότερη. Πάντω, εμεί αυτό που προσπαθούμε είναι να δεσμευτούν όλοι οι εταίροι μας ότι θα υπάρχει διαδρομένος διάλογος με την κοινωνία των πολιτών, του εταίρου και μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες εταίρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθώντας να υπάρχει μια φορά το χρόνο μια κοινή συνάντηση της κοινωνίας των πολιτών. Του χρόνου θα γίνει πρώτη για τις χώρες ΑΤΚ με την ακτή του έχουν δεσμευτεί να κάνουν κάτι αντίστοιχο, μια κοινή πλατφόρμα με τις περιοχές της Ανατολικής Αφρικής, το ΕΣΑ, ε, έχουμε μια μελέτη αντικτύπου και θα οργανώσουμε μίνι συναντήσεις με την κοινωνία των πολιτών. και με την ΕΟΚΕ που οργανώνει και αυτή η τέτοια συναντήση Είναι κάτι που ετοιμάζουμε και θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα διάλογο της κοινωνίας των πολιτών όσο πιο διαδρομένα γίνεται. Θα σταματήσω εδώ στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Σεσίλα, για αυτήν την ε, πολύ διεξοδική παρουσίαση των σχέσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρική. Ε, κυρία Σάρα, πήρε και εσείς πρώτο λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ ε, την Επιτροπή για αυτήν την ε, πολύ λεπτομεριακή παρουσίαση. Ε, θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα. Καταρχήν να πω βέβαια ότι επιχαίρω ιδιαίτερα το γεγονό ότι συζητούμε αυτό το θέμα σήμερα εδώ, αλλά το ζήτημα βέβαια για μα είναι οι πολίτε, οι άνθρωποι τη Αφρική. Δηλαδή, Αναφερθήκατε εδώ σε διάφορες οργανώσεις, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην ε, Αφρική οι οποίοι δεν καταφέρουν να επιβιώσουν. Άρα λοιπόν, ποιε είναι οι επαφές που έχετε με τους ίδιους τους ανθρώπους. Αναφερθήκατε από εκεί και μετά στον αγροτικό ε, τομέα και πράγματι είναι σημαντικό το να υπάρχουν ε, καλύτερες εμπορικές σχέσεις, αλλά πώ ακριβώς παράγονται αυτά τα προϊόντα. Ε, επιβάλλονται οι ίδιοι κανόνες σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την ευημερία των ζώων, την προστασία των ζώων και ούτω καθεξής. Ένα τρίτο σημείο, σε ό,τι αφορά δηλαδή την ε, βιοπικιλότητα δεν υπάρχει εδώ κάποια αποχώρηση τη βιοποικιλότητα. Τι έχετε να πείτε σχέση με αυτό. Ένα ακόμα ζήτημα. Ε, ανάπτυξη και εμπόριο. Ε, ναι, οι βασικέ εμπορικέ σχέσει, ε, αν θέλετε, είναι οι σημαντικότερε ανάμεσα στην Αφρική και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την κατοχή γεών δεν έχει ε, ε, περιέλθει στην κατοχή της Κίνας ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των εδαφών. Ευχαριστώ, Λεπρόεδρος, κύριε Γκουρή. Thank you so much, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν με επιτρέπετε θα χρησιμοποιήσω τη μετρική μου γλώσσα. Ευχαριστώ ε, για ε, την παρουσίαση που ακούσαμε από την εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ε, όλες αυτές τις πληροφορίες οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες. τώρα, στο πλαίσιο της άσκησης εμπορικής πολιτικής που συζητάμε εδώ θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι αλλά και ρεαλιστέ ταυτόχρονα. Θα πρέπει δηλαδή να ε, προωθούμε project ε, τα οποία μπορούν να επιφέρουν απτά αποτελέσματα. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που συζητήσαμε τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουμε για τους κλάδους ε, του χάλιβα και του αλουμινίου, έτσι και εδώ στη σχέση μας με την Αφρική η εμπορική πολιτική δεν μπορεί να επιλύσει όλα τα προβλήματα. Θα πρέπει δηλαδή να επιτύχουμε πρόοδο, αλλά πρόκειται και για μια ήπειρο όπου υπάρχει ε, υποφέρουν πολλοί άνθρωποι και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τους ε, βοηθήσουμε. Δηλαδή ναι, στις δυνατότητες για περισσότερο ελεύθερο εμπόριο, αλλά προς το παρόν νομίζω πως δεν είναι ρεαλιστικό να αναλογιζόμαστε μια πραγματικά συνολική εμπορική συμφωνία ε, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Αφρικής. Υπάρχουν μία σειρά από διαφορετικές συμφωνίες που υφίστανται και τις οποίες μόλις τώρα μας παρουσίασε εκπρόσωπος της Επιτροπής και θεωρώ πως θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτές τις υφιστάμενες συμφωνίες προκειμένου να βοηθήσουμε στο μέγιστο δυνατό της εν λόγω χώρες. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργήσουμε περισσότερο εμπόριο και καλύτερης ποιότητας εμπόριο εάν υποστηρίξουμε τις χώρες της Αφρικής ταυτόχρονα, εάν τις σεβόμαστε αυτές τις χώρες και αν δεν τους υποβάλλουμε υποχρεώσεις τις οποίες δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν ή με τις οποίες δεν μπορούν να συμμορφωθούν. Δηλαδή θα πρέπει να επιβάλλουμε υποχρεώσεις αλλά ταυτόχρονα με τον απαραίτητο σεβασμό και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους. Γιατί αν είμαστε υπερβολικοί τότε αυτό που θα κάνουν λόγω χώρες θα είναι να στραφούν σε άλλους εμπορικούς εταίρους. Και οι τρίτες χώρες δηλαδή οι οποίες ήδη έχουν καταλάβει ένα κομμάτι τη πίτα, αν θέλετε, στην Αφρική, θα καταλάβουν ακόμα μεγαλύτερο με καταστροφικέ συνέπειε για αυτή την Ήπειρο. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε προγράμματα ε, τα οποία θα οδηγήσουν σε πραγματική πρόοδο σε αυτέ τι χώρε σε ό,τι αφορά την παιδεία γενικότερα, δηλαδή την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και ούτω καθεξή. Τομεί δηλαδή στου οποίου θα πρέπει να επενδύσουμε. Και να σα δώσω δύο παραδείγματα. Εάν έχουμε δηλαδή υπερβολικά πολλά μηχανήματα που θα εξαγάγουμε εκεί, χωρίς όμως να συνοδευτούν αυτά από τους κατάλληλα καταρτισμένους τεχνικούς, δεν θα υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα όσο ακριβά και αν είναι αυτά τα μηχανήματα και σε τίποτα δεν θα συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων. Εάν λοιπόν δεν ε, οθετήσουμε την κατάλληλη στάση, τότε θα μπορούσε για παράδειγμα η Κίνα να κατασκευάζει νοσοκομεία ε, στι χώρε τη Αφρική, αλλά όχι χρησιμοποιώντας εργατικό δυναμικό αυτών των χωρών, αλλά με προσωπικό από την ίδια την Κίνα, το οποίο εργάζεται για πάρα πολύ χαμηλά ε, εισοδήματα, πράγμα το οποίο τελικά έχει ανεδικές συνεπίες για τι τοπικέ οικονομίε. Ευχαριστούμε πάντως την Επιτροπή για τις προτάσεις που κάνει και από εκεί και μετά ε, το ζήτημα της μετανάστευσης, το οποίο αποτελεί και απειλή μέσα στην, ε, ε, στην ερχόμενη δεκαετία, θα είναι πιο διαχειρίσιμο αν ακριβώς κατευθύνουμε την παροχή βοήθειας εκεί όπου αυτή είναι απαραίτητη. Ευχαριστώ. Okay. Thank you very much. Um, I am encouraged by the developments... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για την πληρέστατη παρουσίασή σας για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική προς την Αφρική. Σε συνέχεια αυτό που είπε η συναδελφός μας, θέλω και εγώ να ρωτήσω για το μετακοτονού. Πώς έχουν, πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις, ποια σημεία είναι τα δύσκολα στις διαπραγματεύσεις τι κάνετε για να λύσετε τα σημεία αυτά, ποια είναι η συνεργασία σας με την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και τέλος για τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Υπάρχει ουσιαστική ρήτρα και σε αυτήν και σε, στις διμερείς συμφωνίες το θέμα του κλίματος. Κύριος Μπουζουά. Ευχαριστώ σε σχέση με τις προτεραιότητες που αναφέρθηκαν και από τη νέα και από την παλιά επιτροπή, η Αφρική πρέπει να είναι ένας ε, βασικός τέρος μας, είναι γειτόνας και με πολλές δυνατότητες, παρότι έχει και πολλά προβλήματα. Εμείς είμαστε ακόμα πίσω όμως σε διάφορα σημεία θα πρέπει να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία ανάπτυξη. Ξέρουμε όλοι ότι η Κίνα είναι εξαιρετικά δραστήρια στην Αφρική, επενδύει τεράστια κονδύλια στους τομείς που την ενδιαφέρουν, απορροφά πρώτες ύλε, σπάνια προϊόντα που είναι ουσιαστικά για την χώρα. Είναι όμως ουσιαστικά και για μας. Η Ευρώπη εδώ μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχω λοιπόν κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με αυτά που είπε η Επιτροπή. Η Κομισιόν μπορεί να συμβάλλει στην υλοποίηση μιας αφρικανικής ενίας αγοράς. Δεύτερο. στην πολιτική της Ένωσης για την Αφρική, ξέρω, είναι γνωστό ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στην κατάρτιση, την εκπαίδευση. Περιλαμβάνεται στην αναπτυξιακή πολιτική, φαντάζομαι ναι. Μπορεί το εμπόριο λοιπόν να παίξει έναν ρόλο στον τομέα αυτό. Είναι σημαντικό και πρέπει να τονίσουμε ότι ήμουν υπουργό στη Φλάνδρα για ένα μεγάλο διάστημα και ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά που φεύγουν από το σχολείο νέα, μικρά ακόμα, άρα πρέπει να δώσουμε μία έμφαση στην σχολική εκπαίδευση των παιδιών, τη χειραφέτηση των γυναικών για να βοηθήσουμε συνολικά την κοινωνία στην Αφρική. Εκεί είναι η βασική δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Είναι δυνατόν να δώσουμε έμφαση στην ενίσχυση των ε, ικανοτήτων των προσόντων μέσω του εμπορίου. Ξέρω ότι κάποιες επιχειρήσεις έχουν επιφυλάξεις γιατί δεν έχουν επαρκές ε, εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό. Αναφερθήκατε επίσης στη Νότιο Αφρική και σωστά που επηρεάζει τον κλάδο των ε, πουλερικών όχι πάντα θετικά. Θέλω να υπάρχει ταχύτερη δράση της Κομισιόν στον τομέα αυτό όταν διαπιστώνει δηλαδή ε, προβλήματα στη Νότια Αφρική. Οι υπηρεσίες της κυρίας Μάλστρομ είχαν πει ότι σε ένα προηγούμενο επεισόδιο δεν μιλούσαμε για dumping αλλά για ε, μορφές αντίστοιχες με το dumping που θα έπρεπε να αποφεύγονται. Σα Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την Επιτροπή που μας παρουσίασε τις σχέσεις ε, και την εξέλιξή τους κατά τελευταία χρόνια. Ε, κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει συμβεί και θα ήθελα να το αναθέσουμε ως καθήκον στη Νέα Επιτροπή είναι το εξής. Θα πρέπει να χαράξουμε, να ε, δημιουργήσουμε ουσιαστικά μια ε, καθολική εμπορική ε, στρατηγική σε ό,τι αφορά πολύ συγκεκριμένες περιοχές και χώρες, Γιατί συχνά αντιμετωπίζουμε την Αφρική σαν να ήταν μια περιοχή ιδιαίτερα ομοιογενής, πράγμα που δεν ισχύει. Αλλά τι θέλω ακριβώς να πω, να σας το εξηγήσω. Ένα βασικό πρόβλημα που έχουμε σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με την Αφρικανική Ήπειρο και τι διάφορε χώρε τη είναι ότι το επίπεδο των, των εμπορικών συναλλαγών είναι πολύ χαμηλό, γιατί βλέπουμε, για παράδειγμα, πόσο λίγε είναι επιχειρήσει ευρωπαϊκέ οι οποίε ενεργοποιούνται εκεί. Επίση, το επίπεδο των επενδύσεων είναι πάρα πολύ χαμηλό και ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένο. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τι επενδύσει, ε, το ίμιση των επενδύσεων συγκεντρώνεται ε, στην ε, Νότιο Αφρική, τη χώρα δηλαδή, και μετά το υπόλοιπο 40% στι χώρε τη Βορείου Αφρική. Τίποτα δηλαδή στην υποσαχάριο Αφρική. Πράγμα το οποίο καταδεικνύει ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και το οποίο είναι το ότι έχουμε, δεν έχουμε να κάνουμε ε, σε ό,τι αφορά αυτές τις χώρες με ανεπτυγμένες οικονομίες της αγοράς και κατά συνέπεια εκεί δεν βρίσκονται και κατάλληλοι ε, επιχειρηματικοί εταίροι για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ε, πράγμα τι σημαίνει, που, που, τι σημαίνει. Όχι ότι θα πρέπει να αφήσουμε κατά μέρο αυτήν την ε, Ήπειρο, αλλά ότι θα πρέπει να χαράξουμε μια εμπορική στρατηγική με τρόπο για παράδειγμα, που το κάνει και η Κίνα, χωρίς βέβαια να ε, ακολουθούμε τη δική της πολιτική. Δηλαδή τι κάνει. Ε, ε, συνδυάζει πάρα πολύ επιτυχώς την ανθρωπιστική βοήθεια, την εμπορική πολιτική και την επενδυτική πολιτική με πολύ επιτυχημένο λοιπόν τρόπο, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη της την προστασία του κράτους δικαίου, την επεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ούτω καθεξής. Όμως εκείνο που θα πρέπει να ζηλέψουμε το εισαγωγικό από την Κίνα είναι ακριβώς αυτή η στρατηγική προσέγγιση και ο συνδυασμός των πολιτικών Με τις EPAs λοιπόν αυτές συμφωνίε ε, ε, εταιρική ε, σχέση μπορούμε ακριβώ να καταφέρουμε κάτι περισσότερο, γιατί είναι κάτι περισσότερο από εμπορικέ σχέσει. Αλλά ο συνδυασμό με την ανθρωπιστική υποστήριξη, με υποχρεώσει επενδύσεων, με πολύ συγκεκριμένε στοχευμένε προσπάθειε σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την αύξηση του επίπεδου κατάρτιση εκεί, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικό. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ε, υποβοήθηση της ε, ανάπτυξης των ε, υπαίθριων περιοχών, της αγροτικής δηλαδή ανάπτυξης. Άρα λοιπόν αυτό που θα πρέπει να συζητηθεί και με τη Νέα Επιτροπή είναι ακριβώς αυτό. Υπάρχει πρόθεση να κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε πραγματικά μία συνεπή και συνολική καθολική στρατηγική απέναντι σε αυτές τις χώρες ή θέλουμε μια ζωή να έχουμε αποσπασματικές στρατηγικές και μέτρα. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Η Χάιντι Χάουταλα έχει το λόγο. Ναι, ακούσαμε ε, από την Επιτροπή να αναφέρεται και στο ζήτημα των αλυσίδων αξία. Ε, και διαπιστώνουμε ότι τα ε, δάση δεν υφίστανται πυρκαγιέ μόνο στην Αμαζονία, αλλά και για παράδειγμα στι περιοχέ τη Κεντρική Αφρική βλέπουμε πολλέ πυρκαγιέ. Οπότε εμεί ω Ευρωπαίοι καταναλωτέ και ω ευρωπαϊκέ επιχειρήσει ε, είμαστε συνεργοί αν θέλετε, σε αυτό το φαινόμενο, γιατί έχει πολύ συχνά να κάνει με την υφαρπαγή εδαφών, με την αποψήλωση των δασών προκειμένου εκεί να εμποκατασταθούν από ε, αγροτικά προϊόντα τα οποία στη συνέχεια κατευθύνονται προς εξαγωγή και ούτω καθεξής. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ε, μία απροθυμία από την πλευρά για παράδειγμα των ε, παραγωγών κοκοφίνικα σε ό,τι αφορά ακριβώ την, την ευθυγράμμιση με τέτοιου είδου ε, πολιτική και θα ήθελα να ξέρω εάν η νέα Επιτροπή έχει κάποιο σχέδιο προκειμένου ακριβώ να διασφαλίσει διαφάνεια αλλά και ανάληψη των ευθυνών στην αλυσίδα αξία. Ε, γιατί θα πρέπει ε, να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν πάνω από 2 εκατομμύρια παιδιά τα οποία εργάζονται σε τέτοιου είδου εφητείε κοφινίκων στην Αφρική. Άρα λοιπόν αυτό που ανέφερε και η για πρίγμα είναι πολύ σημαντικό ότι δηλαδή βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη συχνά ε, κατάσταση τα παιδιά. Και επίση η αποψήλωση είναι ένα μεγάλο ε, πρόβλημα, ειδικότερα για παράδειγμα σε ό,τι αφορά ε, τα ορυκτά. Σε σχέση με το οποίο, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βάλει υποχρεωτικά μέτρα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο τη αλυσίδα ακριβώ παραγωγή αξία. Τι μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε από τη νέα Επιτροπή. Κάτι ακόμα που είναι σημαντικό είναι το ζήτημα τη διακυβέρνηση, πράγμα το οποίο δεν αναφέρθηκε. Εάν θέλουμε δηλαδή να έχουμε μια επιτυχημένη εταιρική σχέση με τι χώρε τη Αφρική στο μέλλον, θα πρέπει να υπάρχει και χρηστή διακυβέρνηση. Και τι σημαίνει αυτό, ότι χρειαζόμαστε καθαρέ εντό εισαγωγικών ε, οι οποίε είναι υπόλογε στους λαού τη και οι οποίες ε, υπηρετούν ακριβώ τι ε, τις ίδιες τις χώρες και όχι ιδιωτικά συμφέροντα. Yes, thank you very much. And first of all, thanks a lot for this very excellent uh, introduction. Ε, κυρία Βαν θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την Επιτροπή ε, για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, η οποία ήταν έδωσε ταχύτητου σεμιναρίου για τα νέα μέλη εδώ. Εγώ όμω θα ήθελα να θέσω ένα διαφορετικό ερώτημα. Αναφερθήκατε ε, στου λόγου για του οποίου η Αφρική θα πρέπει να αποτελέσει μία από τις προτεραιότητες, αν όχι την απόλυτη προτεραιότητα της Ευρώπης σε ό,τι αφορά ε, την ε, παγκόσμια ανάπτυξη, το εμπόριο και ούτω καθεξής, όπως ε, συμφωνούν και πολλοί συνάδελφοι. Όμως τα ζητήματα της κοινωνικής ανισότητας, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της μετανάστευσης είναι και αυτά ζητήματα που σχετίζονται με την εμπορική πολιτική. Άρα λοιπόν το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής για παράδειγμα και τα ζητήματα της μετανάστευσης θα πρέπει να επιλύονται κατευθυνόμενα όλα προς την ίδια κατεύθυνση. Άρα λοιπόν, ε, σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες εντερική εταιρικής σχέσης, με κατά πόσο θα πρέπει να εξελιχθούν σε κανονικές ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου ε, με τα απαραίτητα κεφάλαια ή όχι. Ε, θεωρώ πως αυτή είναι η οχι θεωρω πως αυτη προσέγγιση, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές ανισότητες και κλιματική αλλαγή. Βλέπουμε να υπάρχουν κεφάλαια τα οποία περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την καθαρή και βιώσιμη παραγωγή ενέργειας. Και εκεί σε στενή συνεργασία με τις αφρικανικές κοινότητες ε, θα πρέπει να τις ε, βοηθήσουμε να περάσουν άμεσα ε, στην εποχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γιατί Εκεί ακριβώς έχουμε να κάνουμε και με τα σχετικά κεφάλαια στις ε, Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου ε, σε ό,τι αφορά ακριβώς την ε, βιώσιμη παραγωγή ενέργειας. Έχουν δηλαδή ασκηθεί κριτικές σε αυτά τα κεφάλαια που περιλαμβάνονται σε λόγω συμφωνίες γιατί θεωρούνται πως είναι αδύνατο να εφαρμοστούν στην πράξη αλλά και δεν έχουν διαδεσμευτικό χαρακτήρα. Εάν λοιπόν θέλουμε να βοηθήσουμε την Αφρική να ανταποκριθεί στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και μάλιστα σε όλες τις παροχές της Αφρικής τότε θα πρέπει πρέπει να ε, μεταρρυθμίσουμε αυτό το κομμάτι της εμπορικής πολιτικής που ασκούμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο Χαλμούτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτήν την ε, παρουσίαση που έγινε από την Επιτροπή ως προς το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ε, κ. Γιούνκερ, είχε αναφερθεί σε μια εταιρική σχέση ε, μεταξύ όμω ομοτήμων. Ε, αυτό τον έφερε το 2018 και θα ήθελα να ακούσω κατά πόσο η νέα επιτροπή είναι διατεθειμένη να ακολουθήσει την ίδια προσέγγιση. Δηλαδή μια ισότιμη εταιρική σχέση. Και ε, εν ώψη ακριβώς της δημιουργίας ε, στο μέλλον μιας ζώνη ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρική στο πλαίσιο των εξελίξεων τώρα ε, βλέπουμε πως έχουμε τρεις επιτρόπους οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι ε, για αυτή, τη δημιουργία αυτή τη ομότιμη εταιρική σχέση. Καταρχήν, είπα του εκπρόσωπο για τι εξωτερικέ σχέσει ε, και μετά ο Επίτροπο για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωή, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Και μετά ο Επίτροπο σε ό,τι αφορά τι διεθνεί εταιρικέ σχέσει. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω ε, στο πλαίσιο της άσκησης εμπορικής πολιτικής θα αναλάβουν αυτόν τον ρόλο οι εν λόγω επίτροποι. Γιατί παλαιότερα οι εν λόγω συμφωνίες EPA αφορούσαν επιμέρους περιοχές. Οπότε ε, υπάρχουν διαφορετικές ε, χώρες για παράδειγμα οι οποίες εξελίσσονται με διαφορετικό τρόπο όπως για παράδειγμα η Γκάνα, η Ακτή του Ελεφαντοστού, η Κένια. Για αυτέ λοιπόν τις χώρες, στο πλαίσιο των οποίων δηλαδή έχουν λειτουργήσει οι EPA, θα ήταν κάτι χρήσιμο το να περάσουμε ε, από τι EPA τώρα προ τι FTA που θα αφορούν το σύνολο τη ε, Αφρικανική περιοχή. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν συμφωνώ με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι σε ό,τι αφορά ε, την επίτευξη των διάφορων στόχων, σε ό,τι αφορά την προώθηση δηλαδή τη υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν ε, διαρωτώ κατά πόσο, ε, ε, ποιες μάλλον θα είναι επιπτώσεις ε, στις επιμέρους οικονομίες αυτών των χωρών στο πλαίσιο εφαρμογής αιτίων συμφωνιών. Και αν λάβω υπόψη μου αυτά τα επιχειρησιακά εργαλεία τα οποία προβλέπονται στις νέες FTA, για παράδειγμα με την προστασία των κανόνων, των κανόνων καταγωγής και την κατάργηση των εμπορικών εμποδίων κατά το 90%, έτσι ώστε κατά 90% να έχουμε δημιουργήσει ακριβώς μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου, τότε λοιπόν τίθεται το ερώτημα κατά πόσο εμείς από την δική μας πλευρά θέτουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις έτσι ώστε με τη σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας θα υποστηρίξουμε τη βιομηχανική ανάπτυξη εκεί. Για παράδειγμα υπάρχουν συμφωνίες διευκόλυνσης του εμπορίου στο πλαίσιο του ΠΟΕ και ούτω καθεξής, αλλά ποιες είναι, ποια είναι τα συμπληρωματικά μέτρα και τα ε, εξατομικευμένα προγράμματα τα οποία μπορούν να προωθήσουν ακριβώς αυτή την αυξημένη οικονομική αυτονομία των ε, αφρικανικών χωρών. Αυτό είναι σημαντικό και εκεί θα έρθει και το benchmark ε, του 2030, στο πλαίσιο του οποίου και εμείς και οι αφρικανικές χώρες θα πρέπει να και να δούμε κατά πόσο έχουμε προχωρήσει σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ατζέντα ε, των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Και σε αυτό λοιπόν το επίπεδο θα πρέπει να ε, παράσχω υποστήριξη για την ε, πλήρωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στις αφρικανικές ε, χώρες και βέβαια είναι ε, πολύ σημαντικό το γεγονός που ανέφερε η εκπρόσωπος της Επιτροπής ότι θα έχουμε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους, ε, δις, ανθρώπους οι οποίοι θα ζουν στην Αφρική το 2050. Ευχαριστώ. Κοκοφίνικας. Το έθεσε κάποιος ε, βουλευτής. Σε σχέση με την παιδική εργασία, την μείωση του, των δασών κλπ. Στη Δυτική Αφρική είναι το θέμα. Γκάνα, κτήλε, ελεφαντοστού και γκαμπών είναι 70% των εξαγωγών κοκοφίνικα στην Ένωση. Άρα εκεί έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε. Είμαστε μεγάλοι πελάτες και υπάρχουν και προβλήματα ιδίως στην ε, ακτήρα για τα θέματα της παιδικής εργασίας ε, το θέμα επίσης της αποψήλωσης των δασών ε, και της ε, φύτευσης κοκοφινίκων είναι ένα άλλο ζήτημα. Το έχουμε συζητήσει και με την κυβέρνηση της Ακτής Εφαντοστού και με τον κλάδο για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να επιβάλλουμε απομονωμένα. Πρέπει να έχουμε ένα διάλογο με την κυβέρνηση, τους επιχειρηματίες, για να βρούμε κάποιες λύσεις, γιατί το θέμα είναι δύσκολο που θα αλλάξει την πρακτική, ουσιαστικά για την κυβέρνηση. Ε, και δεν θέλουμε κάτι να μην εφαρμοστεί εν τέλει. Το παρακολουθούμε προσπαθώντας να βρούμε μία λύση. Την άλλη ή την παράλληλη εβδομάδα οργανώνεται από την αντιπροσωπεία μας ένα εργαστήρι για το θέμα αυτό στην ακτή Ελεφαντοστού. Συνεργαζόμαστε και με του, τις οργανώσεις κακαοπαραγωγών και θα δούμε πώς είναι οι εναλλακτικές. Επίσης, ε, η Εφημερία των ζώων, κάποιος το έθεσε, είναι σημαντικό ε, να παρακολουθούμε το πώς γίνονται οι εξαγωγές από την Αφρική σε μας. Πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας. Οι συμφωνίες μας δεν περιλαμβάνουν το θέμα της ευημερίας των ζώων αυτό καθεαυτό, αλλά στις συμφωνίες ESA που ξεκινούμε τώρα θα συμπεριλαμβάνουμε και την συνεργασία στον τομέα. Πρόκειται για έναν τομέα που έχουμε συζητήσει για το πώς ενισχύσουμε την ε, συνεργασία στον τομέα αυτό. Δυτική Αφρική, τι γίνεται με την Ιγυρία. δεν έδωσε κάποιο μήνυμα ότι θέλουν να υπογράψουν την Περιφερειακή Συμφωνία. Το συζητούμε μαζί τους. Είμαστε ανοιχτοί στις συζητήσεις αν έχουν προβλήματα με την υφιστάμενη. Προτιμούμε προφανώς να υπάρχει μια περιφερειακή, όχι ε, ε, διμερή συμφωνία, αλλά πρέπει να συζητηθεί με όλες τις χώρες. Ε, άμα τώρα το μπλοκάρει η Νιγηρία δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Η Νιγηρία έχει υπογράψει μια VFCFT, τελευταία χώρα ήταν. Θα δούμε αν υπάρχει κίνηση προς αυτό. Δεν εξαρτάται από μας. Περιμένουμε να δούμε τι, θα θέλει να κάνει η κυβέρνηση της Νιγηρίας. Ζάμπια. Γιατί δεν υπογράψαμε ESA. Μπορώ να σας πω ότι ήταν συμβαλόμενο μέρος στην συμφωνία του ESA, δεν το υπέγραψαν εν τέλει, γιατί ήθελαν να συμπεριληφθούν περισσότεροι τομεί στην EPA, όχι μόνο εμπόριο αγαθών, που σημαίνει ότι Ε, έχουν άλλα ενδιαφέροντα και άλλα συμφέροντα. Θέλουν τώρα να μπουν, ξαναρχίσαμε να συζητούμε, αυτό είναι καλά νέα, τους είπαμε τι πρέπει να κάνουν. Απλώς πρέπει να το υπογράψουν και να ξεκινήσει η διαδικασία της κύρωση. Ιδίω γιατί διαπραγματευόμαστε περισσότερα σημεία, οπότε πρέπει να παρακολουθούν τις συζητήσεις. ε, απώλεια εσόδων λόγω υποτίμησης και μείωσης των ε, δασμών με τις αφρικανικές χώρες. Αυτό το συζητούμε με τους εταίρους της... Ε, συνήθως έχουμε μελέτες για κάθε χώρα να δούμε τι απώλειες υπάρχουν, πώς μπορούμε να τις υποστηρίξουμε για να προσαρμόζονται στην απώλεια εισοδήματος που θα έχουν από το γεγονός ότι δεν θα εισπράττουν δασμούς αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι η απελευθέρωση γίνεται βαθμιαία. Τον πρώτο χρόνο απελευθερώνουμε μικρά προϊόντα, τα περισσότερα απελευθερώνονται στο τέλος της διαδικασίας, στα 15-20 χρόνια ανάλογα με την EPA. Η διαδικασία είναι μακρά, δεν αλλάζει η, το, φο, το ποσοστό ε, ξαφνικά. Ο αντίκτυπος δηλαδή είναι σχετικά περιορισμένος, μπορούμε να βρούμε τα καταλληλότερα εργαλεία για να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις και τα κράτη. Αυτό επίσης τους βοηθά να προσαρμόσουν και τις απαιτήσεις της κοινωνίας, οπότε γενικά είναι θετικό για τις αλλαγές που μπορούν να κάνουν. Νομίζω ότι κάλυψα. Α, Κίνα. Ναι. Κάποιοι βουλευτές το έφεσαν. Όντως, η Κίνα για, θεωρεί προτεραιότητά της την Αφρική και πολιτικά και οικονομικά. Επενδύουν πολλά. Αν δείτε την ανάπτυξη των επενδύσεων εκεί, προφανώς η πορεία της ανάπτυξης των επενδύσεων της Κίνας είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δική μας, αλλά εμείς είμαστε ακόμα συνολικά πιο πάνω. Ανεβαίνει, υπάρχει ανωδική λοιπόν πορεία, αλλά μην το δείτε ως ε, αρνητικό γιατί παίζουν κομβικό ρόλο στις υποδομές, ε, στην ανάπτυξη των υποδομών εκεί. Προφανώς δεν ακολουθούν τα ίδια στάνταρτ που θα θέλαμε εμείς πάντα. Ή αυτά που θα επιβάλαμε σε μια ευρωπαϊκή εταιρεία. Και οι όροι δεν είναι αυτοί που θα θέλαμε. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι αυτή. Εμείς συζητούμε με την Κίνα για να έχουμε μια περισσότερο κοινή στρατηγική που έχουμε κοινά συμφέροντα, τι μπορούμε να κάνουμε με πιο βιώσιμο τρόπο. Δεν πρέπει δηλαδή να βλέπουμε ότι οι Κινέζοι και εμείς είμαστε μόνο ανταγωνιστές. Νομίζω ότι κάλυψα τις περισσότερες ερωτήσεις. Αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, εδώ είμαι. Ωραιότατα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε για αυτή την ενημέρωσή σα, για τη συζήτηση που κάναμε σε ό,τι αφορά την εμπορική πολιτική σε σχέση με την Αφρική. Κλείνουμε λοιπόν εδώ με την πρωινή συνεδρίαση και στις 3 η ώρα θα ξαναρχίσουμε εδώ και πάλι. Σας ευχαριστώ.